Εντάξει, δεν είμαστε πολυπληθείς, αλλά είμαστε εκλεκτοί. Γιατί έπρεπε να γίνει και μια συνάντηση για τα δύο νομοθετήματα παράλληλα. Αυτοί όμως που είμαστε εδώ πέρα νομίζω θα περάσουμε άριστα. Σας, μπορώ να σας ζητήσω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ε, έχουμε μόλις τελειώσει τη συνεδρία των συντονιστών. Και έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Πρώτα απ' όλα, αύριο δεν έχουμε συνεδρίαση. Επειδή θα αναβληθεί και η ψηφοφορία για τα στεγαστικά δάνεια, έχουμε μία συνάντηση με τον Τόμας Φάιτσερ, τον πρόεδρο της CFC στις 8 Μαΐου αύριο 2 με 3 το απόγευμα λοιπόν. Είσαστε προσκεκλημένοι. Και αν χρειάζεται να σας το υπενθυμίσω, η EFC, δηλαδή η Οικονομική και Χρηματοπιστωτική ε, Επιτροπή, είναι επιφορτισμένη με το να προετοιμάζει τις ε, συνεδριάσεις του ΕΚΟΦΗΝ και να παρακολουθεί την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση στα κράτη-μέλη, δίδοντας τακτικές εκθέσεις στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Ιδιαίτερα η Επιτροπή αυτή, η EFC, παίζει σημαντικό ρόλο στην συνεχιζόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας να συζητήσουμε θέματα αυτά, αυτά τα θέματα, ιδίως διαδικασίες για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλημάτων. Θα είναι μια ανοιχτή συνεδρία συντονιστών, χωρίς ε, μέσα ενημέρωσης, χωρίς ε, μετάδοση στο διαδίκτυο. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια πλήρη ανταλλαγή απόψεων. Επίσης έχουν λήξει οι διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Επεκτείνεται με τις τροπολογίες αυτές <clears throat> και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο η σφαίρα εφαρμογής αυτής της τράπεζας. Είναι μια επαναδιαβούλευση με την Επιτροπή μας. Είχαμε ένα τριγωνικό διάλογο που έλαβε χώρα στις 24 Απριλίου καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία και υπήρξαν κάποιε λεπτομέρειε οι οποίε διευκρινίστηκαν σε μια μεταγενέστερη γραπτή διαδικασία μεταξύ των διαπραγματευτών. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι βάσει του άρθρου 70 παράγραφος 3 να ζητήσω τη διαβούλευση με την Επιτροπή μας. Αν κάποιος σκιώδης εισηγητής θέλει να μιλήσει ας το κάνει τώρα. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις το τροποποιημένο κείμενο θα πάει στην Ολομέλεια και τον Ιούνιο θα γίνει ψηφοφορία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Καμία. Ωραία. Οπότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προδιέγραψα. Κόφι, παρακαλώ. Choose moment to come with coffee. Έρχονται πια πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή να, να μας ε, σερβίρουν καφέ, διότι τώρα προχωρούμε σε ανταλλαγή απόψεων με τον Βάλτερ Ράντερμαχερ, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωστάτ, με μεγάλη χαρά χαιρετίζω τον Βάλτερ στην Επιτροπή μας. Είμαι σίγουρη θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην αρχή θα κάνω μια μικρή εισηγήση. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά προσέρχομαι ενώπιόν σας για να ανταλλάξουμε απόψεις για ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, πώς έχουν τα πράγματα και τι στρατηγικές προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Η σημερινή ακρόαση είναι πρώτη φορά που διοργανώνεται για να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να γίνει και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο μια δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό για να μπορέσουμε έτσι να εξυγχρονίσουμε τα στατιστικά μας συστήματα η Κομισιόν ζήτησε σκληρά μέτρα που είναι απαραίτητα. Και η δική σας υποστήριξη είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες και οι διαχειριστικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Τώρα όλοι δέχονται ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι fit for purpose, αξιόπιστα και να αποτελούν τμήρμα της λύσης και όχι του προβλήματος για να διευκολύνουν, να προωθούν τη δημοκρατική νομιμότητα. Στατιστικά στοιχεία καλής ποιότητας ανέκαθεν ήταν, βρίσκονταν στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και είναι από τα κυριότερα τμήματα της Κομισιόν. Από το 1957 ήδη έχει οργανωθεί και επειδή τον Ιούνιο θα γιορτάσω τα 60 μου γενέθλια, με περηφάνεια μπορώ να σας πω ότι θα είμαι τρεις μήνες γυρεότερος από το Eurostat που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 52. Εγώ κερδίζω λοιπόν. Λοιπόν, η στατιστική μας υπηρεσία έχει ε, πολύ εξελιχθεί με βάση ένα κοινό σύστημα παραγωγής ή υποβολής των στοιχείων σε συνεργασία με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Μέχρι πρόσφατα αυτό το σύστημα δούλευε καλά. Τα στατιστικά μας στοιχεία πάντοτε έγκαιρα υποβάλλονταν και υποβοηθούσαν την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Από την ΕΚΑΧ ήδη, το 57 σας είπα, Uh, λοιπόν, τώρα από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ε, δημιουργήθηκαν άρχισαν να δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα γιατί υπάρχουν νέα αιτήματα, νέες ανάγκες για στατιστικά στοιχεία με βάση τις κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές και άλλες καινούργιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Δεύτερον, οι στατιστικές υπηρεσίες δεν έχουν πολλούς πόρους. Δηλαδή, μεγαλύτερη ζήτηση αλλά λιγότερη πόρη. Και περισσότερη ευθύνη απαιτείται. Οι πολιτικές και νομικές αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται ημιαυτόματα για την ερμηνεία των ποσοτικών στοιχείων δεν υπάρχουν ακόμη. Δηλαδή, οι στατιστικοί θεωρούνταν ως ένα πρώτο βήμα για τη λήψη αποφάσεων, αλλά τώρα αυτοματοποιείται όλο και περισσότερο. Μεταξύ δικτών και αποφάσεων υπάρχει πολύ μεγαλύτερη και αυτόματη σχέση πια. Τρίτον, δυστυχώς τελευταία ορισμένα ατυχή γεγονότα που όλοι τα ξέρετε δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε ανεξάρτητα και αξιόπιστα στοιχεία, επίσημα στοιχεία. Αυτές είναι οι προκλήσεις που δεν μπορούμε να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε. Κυρίες και κύριοι, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές με την Ευρώπη. Ευρωπαϊκή λύση στο στατιστικό πρόβλημα για να είμαστε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε το στίχημα της αποτελεσματικότητας με μεγαλύτερη συνεργασία και λιγότερες επικαλύψεις. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι θα δημιουργηθεί ένα πραγματικά ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες και πολλές νομικές μεταρρυθμίσεις. Θα αναφέρω κυρίως το 2009 ο λεγόμενος στατιστικός νόμος δηλαδή ο κανονισμός 223 εγκρίθηκε. Η ενεργότατη συμβολή σας εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και από εμά γιατί χρειάζεται όντως πολύ αυστηρότερος ορισμός των προτύπων ποιότητος και συλλογής των στοιχείων. Στον λίγο χρόνο από τότε μέχρι σήμερα το στατιστικό αυτό νομοθέτημα αποδείχτηκε πολύτιμο. Τον ίδιο χρόνο μάθαμε ότι σε μία χώρα μέλος στην Ελλάδα δηλαδή υποβάλλονταν αναλυθή στοιχεία. Τον Ιανουάριο του 10 υποβάλαμε σε μεγάλη λεπτομέρεια το βαθμό και το ποσότητα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Ελλάδα από στατιστικής σκοπιάς και επίσης μάθαμε και άλλα ατυχή μαθήματα, άλλα αρνητικά μαθήματα, ότι τα προβλήματα σε μία χώρα μέλος μπορούν να υπονομεύσουν το σύνολο της στατιστικής υπηρεσίας της Ένωσης. Και έτσι πολλαπλασιάστηκαν οι πολλαπλές δημοσιονομικές κρίσεις και οι κρίσεις χρέους. Και έτσι. Πρέπει να ξεριζώσουμε τέτοιες, τέτοια προβλήματα από τη ρίζα τους σε συνεννόηση με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος πρέπει να γίνουν θεσμικές μεταρρυθμίσεις, να αυξηθεί η ποιότητα των στοιχείων και να επανέλθει η Ελλάς στον σωστό στατιστικό δρόμο. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λοιπόν, από τον Απρίλιο, από τις 23 Απριλίου, για τέταρτη φορά δημοσιεύουμε τα στοιχεία τα στοιχεία για τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Επίσης πήραμε μαθήματα. Προσπαθούμε πιο πολύ να εγγυόμεθα την ποιότητα των στοιχείων μας, να επαληθεύουμε και να εποπτεύουμε από την αρχή την υποβολή των στατιστικών στοιχείων. Επίσης το, ε, αποκτήσαμε καινούργιες δικαιοδοσίες δημοσιονομικού ελέγχου και τις χρησιμοποιούμε με μεγάλη φρόνηση για να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Παραδείγματο χάρη, τι αιτήσει σας ζητούμε συστηματικότερη συλλογή στοιχείων για προβληματικές και οριακές περιπτώσεις. Δηλαδή θέλουμε να βελτιωθούν όλες οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες στα κριτήρια του λεγόμενου ύψος, του ύψους. Το 9 επίσης η Κομισιόν ενέκρινε μία ανακοίνωση με τίτλο «Ο τρόπος παραγωγής των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων το όραμα της επόμενης δεκαετίας». Και με βάση αυτή την ανακοίνωση συγγράφτηκε ολόκληρο πρόγραμμα εργασίας δικό μας που αντιπροσωπεύει πολύ σημαντική συστημική αλλαγή για όλους τους συνεργάτες μας των στατιστικών υπηρεσιών για καλύτερη διαχείριση των πόρων που διαθέτουμε. Δύσκολο πράγμα, γιατί σημαίνει ότι αλλάζει η νομική αρχιτεκτονική που βασιζόταν σε περίπου 350 κανονισμούς και μας επέτρεπε να συλλέγουμε από πολλαπλές πηγές στατιστικά στοιχεία χωρίς επικαλύψεις, με συνέργειες και με μεγαλύτερη ευελιξία. Έχουμε όμως και ορισμένους φραγμούς που αντιμετωπίζουμε, παραδείγματο χάρη τον βαθμό συνειδητοποίηση την ε, δυσπιστία των χωρών μελών που δεν ε, μας υποβάλλουν τα στοιχεία τους ασμένος και ο δισταγμός τους να εφαρμόσουν μια πιο ευέλικτη μέθοδο με χρησιμοποίηση, πληρέστερη χρησιμοποίηση όλων των δευτερογενών νομικών εργαλείων που διαθέτουμε, ιδιαίτερα των κατά... E Finally, we are... κατεξουσιοδότηση πράξεων. Είναι όμως απαραίτητο καταρχήν να κάνουμε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας και να δούμε πώς θα απελευθερώσουμε ό,τι πόρους διαθέτουμε αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα της ε, πολύ γρήγορης αλλαγής των καταστάσεων που πρέπει να επιτηρούμε. Όπως καταλαβαίνετε μόνο αν είναι υψηλής ποιότητας οι επίσημες στατιστικές έχουν κάποιο νόημα. Και οι ίδιοι θεωρήσατε αυτό το στοιχείο ως ακρογωνιαίο λίθο της νέας τύπου διακυβέρνησης, governance δηλαδή. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα προβλέπεται επισήμως από την εξάμετρο. Εμείς αυτό το δεχόμαστε με χαρά. Να αλλάξει δηλαδή ο στατιστικό, ισχύον στατιστικός νόμος, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, συνεργασία, πρόσβαση σε διοικητικές πηγές και υποχρεωτική χορήγηση εμπιστευτικών μέχρι τώρα στοιχείων με κάποιο είδους συμβόλαιο μεταξύ Κομισιών και κράτους μέλους ώστε όλες οι χώρες μέλη στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο να μετατρέψουν, να μεταφέρουν την νομοθεσία αυτή επιτόπου. Προσβλέπω στις συμβουλές και τις παρατηρήσεις σας γιατί νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι πολύ απαιτητική ως προς τις διαπραγματεύσεις της συναπόφασης ετοιμαζόμαστε να αναθεωρήσουμε το ρόλο του Eurostat για να μπορούμε να αντικατοπτρίζουμε καλύτερα αυτά που απαιτούμε και από τα κράτη-μέλη. Από την εμπειρία μας από το EDP είδαμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη εξισορρόπηση των μακροοικονομικών στοιχείων σε συνδυασμό με την στρατηγική του 2020. Θέλουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και πρότυπα. Τώρα τελειώνουμε την δεύτερη εξέτασή μας της πιθανότητας στατιστικών κυρώσεων στα πλαίσια της εξαμέτρου. Και προσπαθούμε να παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις νέες εξελίξεις για την governance, όπως και την δίμετρο. Και Όλα αυτά επηρεάζουν και τις επίσημες στατιστικές. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η governance. Προτείνουμε μεταρρυθμίσεις και στον προγραμματισμό μας. 13 με 17 έχουμε προβλέψει να εφαρμοστεί το ΕΖΑ, ε, το ΕΖΑ 2010. Ελπίζω τελικά να καταλήξουν όλα αυτά στην εφαρμογή των υψηλοτάτων προτύπων που είχαμε αρχικά προτείνει. Θα υπάρξουν όμως και άλλες προτάσεις, παραδείγματος χάρη. Νέα στατιστική για την ενιαία αγορά. Αυτό είναι καινούριο. Το Simpstat που λέμε εμείς. Να αντικατασταθεί δηλαδή το Intrastat με ένα πολύ πιο απλοποιημένο σύστημα επισήμων στοιχείων για το εσωτερικό εμπόριο αυτό θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά στο να μειωθεί το άχθος της συλλογής στατιστικών στοιχείων. Εν τέλει, η Eurostat, τα ευρωπαϊκά στατιστικά γραφεία εξακολουθούν να εργάζονται για το μέλλον της ευρωπαϊκής στατιστικής, ιδίως μέσα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ΑΕΠ και επέκεινα του 2007, έχουμε δημιουργήσει ένα οδικό χάρτη για να μπορέσουμε να συλλέξουμε οικονομικές στατιστικές που να συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, οι ευρωπαϊκές στατιστικές έχουν περάσει σημαντικές μεταλλαγές τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούσαμε να πράξουμε άλλος. Είμαι έτοιμο να τονίσω τη σημασία του να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος με μια νέα και ε, προδημιουργική πολιτική θα μπορέσουμε να φτιάξουμε το κατάλληλο περιβάλλον για τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurostat θα συνεχίσουν αυτό το εγχείρημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είμαστε μόνοι μας. Η υποστήριξή σας ήταν μια πραγματική βοήθεια για όλα αυτά. Πιστεύω ότι έτσι θα πρέπει να παραμείνουμε στεναροί για τις πολιτικές μας προσπάθειες να καταλήξουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσουμε ότι θα ανταποκριθούμε από αυτά τα οποία, σε αυτά που ζητούν οι πολίτες από μας. Δεν μας φτάνει το status quo. Έχουμε ένα σκληρό αγώνα. Πιστεύω όμως ότι είναι ένας αγώνας για καλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Προσβλέπω στο να έχουμε και πάλι την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε μαζί, να μοιραστούμε πληροφορίες που θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του πώς συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα στην ευκυβερνησία και στην καλύτερη χάραξη της πολιτικής στην Ευρώπη σε ένα ρευστό κόσμο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Walter. Ευχαριστώ, Walter. Η Επιτροπή μας είναι φίλη σου και σαν φίλοι προσπαθήσαμε να σας δώσουμε και περισσότερες αρμοδιότητες. Έχουμε μία μακρά διαδικασία ακολουθήσει, ήδη πριν γίνω εγώ πρόεδρος. Και χαίρομαι που τουλάχιστον σε κάποιους τομείς μπορέσαμε να βοηθήσουμε στα πλαίσια της εξαπλής πρότασης. Τώρα θα έλθω σε ερωτήσεις. Ποιος θέλει να θέσει ερωτήσεις. Ίσως πρώτα να πάρουν το λόγο οι συντονιστές, εφόσον το επιθυμούν βέβαια. Σφέν, έχει ζητήσει το λόγο. Ναι. Κοιτάξτε, ακολουθήστε τη σειρά. Όποιος ζητάει το λόγο, δώστε του το λόγο. Καταρχάς να καλωσορίσω τον κύριο Ράντερ Μάχερ. Νομίζω ότι στα πλαίσια της στατιστικής, των στατιστικών μάλλον γενικότερα υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι είναι σημαντικοί. Το ένα είναι το έλλειμμα και το άλλο είναι το χρέος. Πρόκειται για, για στατιστικούς δείκτες οι οποίες ε, θα έλεγα, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι σημαντικότατοι για τη συγκεκριμένη χώρα που αναφέρατε, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες με τον ένα τρόπο ή τον άλλο έχουν συνεισφέρει στην ε, λιγότερο επακριβή αναφορά των δικτών. Και αυτό μάλιστα συμβαίνει και σήμερα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι μέχρι τη φάση που θα φτάσουμε σε ένα εναρμονισμένο λογιστικό σύστημα όπως ακριβώς και στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς και έχουμε τον DSA και το σύστημα από το 2010, αλλά υπάρχουν προς το παρόν χώρες οι οποίες έχουν σύστημα ισροών ρευστών, άλλες οι οποίες έχουν αναλογιστικό σύστημα και ακόμα και αν όταν όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο μεταφραστούν όταν παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούν θα έλεγα παρερμηνίες και προκαλούν γενικότερα θέματα και όλα αυτά θα τα θα τα χαρακτήριζα θα έλεγα εφάνταστα λογιστικά συστήματα, κάτι το οποίο ε, δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί. Μπορείτε να μας το πείτε αυτό. Λοιπόν, η ερώτησή μου, η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει να αντισταθμίσουμε τη μη ύπαρξη ακριβώς αυτού του συστήματος ε, λογιστικού βάση καταβεβλημένων σε όλα τα κράτη-μέλη, έχοντας την δυνατότητα να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της αλλαγής από το μακροοικονομικό επίπεδο, από το επίπεδο της ισροής, ε, και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν. Αλλά θα ήταν προφανώς πάρα πολύ καλύτερα αν τα κοινά μπορούσαν να καλυφθούν και σε επίπεδο μικρολογιστικό και να έχουμε ένα σύστημα επί τη βάση των καταβεβλημένων ποσών το οποίο να είναι ισότιμο για όλες τις χώρες. Βέβαια υπάρχουν αντιρρήσεις για την εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος. Υπάρχει σκεπτικισμός γιατί το κόστος αυτού του συστήματος σαν παράδειγμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο υποστηρίζουν ορισμένοι το αποτέλεσμα της βελτίωσης την οποία μπορεί να έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τις ε, μελέτες τις οποίες κάνουμε, να κάνουμε μια σωστή σύγκριση των μελετών αυτών στο τέλος του χρόνου και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης τελικά για τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσουμε αυτό το σύστημα. Πάντως δεν θα είναι καθόλου εύκολη η διαδικασία γιατί αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ανησυχίες, ότι το σύστημα αυτό κοστίζει πολύ, το σύστημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για τον δημόσιο τομέα και μάλιστα να πω εδώ ότι οι κοινοβουλευτικοί και σε διάφορες χώρες μέλη διαμαρτύρονται για αυτή την πρόταση και διστάζουν να περάσουν σε ένα τέτοιο σύστημα λογιστικό επί τη βάση των καταβεβλημένων ή δουλευμένων αν θέλετε γιατί ανήκει σε ένα σύστημα διαφάνειας το οποίο ακόμα θα πρέπει να μάθουν να εργάζονται. Πράγματι είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς τη διαφάνεια, λέει η Πρόεδρος. Κλίντς. Σε ευχαριστώ Σάρων, σε ευχαριστώ Βάλτερ για την παρουσίαση εδώ και την προθυμία σου να έχουμε ένα διάλογο. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σχετικά θετικά. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστούν άλλα 60 χρόνια για να μπορέσουμε όλοι να δώσουμε τις ε, απαραίτητες ευρωπαϊκές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εγώ διαπιστώνω ότι οι εμπειρίες μας στο παρελθόν ήταν βέβαια αρκετά αρνητικές μερικές φορές. Είμαι από το 2004 στο Κοινοβούλιο και από το 2005 είχαμε πει ότι το, η Ευρωστάτη παίζει σημαντικό ρόλο στα οικονομικά θέματα, υπήρχε τότε η κατάσταση με τα στοιχεία της Ευρώπης. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρξαν κράτη-μέλη όπως η Γερμανία που έχουν ζητήσει να υπάρχουν περισσότερες αρμοδιότητες στην Eurostat. Και σε αυτά που είπε ο κύριος ε, Σιγκούνα, εγώ είχα ε, εξασφαλίσει να υπάρξει μια καλύτερη μορφή ελέγχου για το λεγόμενο ντοπάρισμα των ε, οικονομικών. Ε, όταν δηλαδή μακιγιάρουν τα κρατήδια ή οι χώρες τα στατιστικά στοιχεία. Και τόνισε ότι αυτό έπρεπε να ξεπεραστεί. Το ερώτημα μου τώρα είναι το εξής. Αν σήμερα κοιτάξουμε παρά όλες τις προέ... Αν κοιτάξουμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Είσαστε σίγουρο ότι συγκρίνουμε μήλα με μήλα και όχι μήλα με ερήφια ή Αμνού με αχλάδια. Είναι σίγουρο ότι έχουμε μια συγκρισιμότητα στα, στα, στα στοιχεία που συλλέγεται. Εγώ ξέρω ότι ακόμα και μέσα σε μια χώρα, μέσα στη Γερμανία παραδείγματο χάρη, τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής χάρη του γερμανικού κράτους για τα θέματα εργασίας είναι διαφορετικά από τα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας στο Βισμπάντε. Δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν και μεταξύ κρατών υπάρχουν διαφορές. Παραδείγματο χάρη, οι εξαγωγέ τη Γερμανία προ Γερμαν... προς τη Γαλλία δεν είναι ακριβώ ίδιε με αυτά που καταγράφεται στη Γαλλία ω εισαγωγέ από την Γερμανία. Γι' αυτό αναρωτιέμαι κατά πόσον είμαστε σε θέση να πούμε ότι μπορούμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Η στατιστική βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα εργαλείο για τους λήπτες απόφασης. Και επομένως δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η στατιστική είναι ένα φετίχ. Όταν μιλάμε για την διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να βλέπω τις στατιστικές σας σαν ένα είδος κλεφτοφάναρου ή ένα είδος φάρου που διαφωτίζει καλύτερα τα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι λήπτες αποφάσεων. Αυτό που λέτε για τη δέσμευση για να δημιουργήσετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, βεβαίω όλα αυτά είναι πολύ καλά. Μπορεί πάντα κανεί να δεσμεύεται για το δημοσιονομικό σύμφωνο, για την ανάπτυξη κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά εμένα δεν με νοιάζει τόσο πολύ η εμπιστοσύνη όσο το να έχουμε επακριβή στοιχεία στατιστικά. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη συγκρισιμότητα των δημοσιονομικών στοιχείων. Έχουμε φτάσει ένα επίπεδο συγκρισιμότητας το οποίο θα έλεγα ότι είναι μοναδικό πλέον. για τα, κριτήρια του, για τα κριτήρια του Μάστριχτ, για το χρέος και το έλλειμμα. Έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία ανάμεσα σε χώρες, οι οποίες ε, δεν συγκρίνονται με τη δικά μας δεδομένα, με τα αμερικανικά δεδομένα, με τα αυστραλιανά δεδομένα, με τα δεδομένα της ομάδας των 20. Έχουμε όμως εδώ ένα σύστημα το οποίο μπορεί να διασφαλίσει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην στατιστική κοινότητα ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Βέβαια το να επιβάλλει κανείς ένα τέτοιο ποιοτικό σύστημα σε όλα τα στατιστικά συστήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σχετικά σαν παράδειγμα με τις υδατοκαλλιέργειες. Να σας δώσω το παράδειγμα των υδατοκαλλιεργειών. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ε, μια διαφοροποίηση γιατί τα οστρακοειδή τα οποία προσμετρώνται στην Γαλλία ή στην Ισπανία ανήκουν σε διαφορετικά μεγέθη από ό,τι σε άλλες χώρες. Σε επίπεδο στατιστικής δηλαδή θα φτάσουμε στην λεγόμενη αρχή των Ηνωμένων Εθνών fitness for purpose. Για ποιο λόγο θέλουμε να διασφαλίσουμε τη, τη συγκρισιμότητα και ποια ποσοστά λάθους μπορούμε να έχουμε ανεκτά. Γιατί είναι σαφές ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι ένα επιπλέον βάρος διοικητικό και είναι και οικονομικό επιπλέον βάρος. Δεν είναι τίποτα δωρεάν. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί σας και να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς ένα από τα συστήματα τα δυνατά στατιστικών μπορεί να εξυπηρετήσει έτσι ώστε να φτιάξουμε όσο πιο κοντά στις ανάγκες σας αυτό το σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Αναφερθήκατε στις συντάξεις, στα συνταξιοδοτικά. Εδώ να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνεται στα στάνταρ των Ηνωμένων Εθνών. Με ένα ενιαίο μέσο δηλαδή μπορούμε εμείς να καλύψουμε το ε, το κρυφό κόστος αν θέλετε, χρέος το οποίο αφορά ε, τα συνταξιοδοτικά. Αυτή είναι η πρότασή μας. Υπάρχουν βέβαια τρεις χώρες οι οποίες σε αυτή τη φάση, στα πλαίσια του ΕΖΑ 2010, θέλουν να μπλοκάρουν το σύστημα και είναι μάλιστα οι τρεις μεγαλύτερες χώρες αυτές. Είδαν ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι αλλά πιστεύω ότι σε συνεργασία με εσά και σε συνεργασία με την Προεδρία έχω την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε έτσι ώστε το σύστημά μας αυτό να περάσει και να έχουμε την πρόπτικη έτσι ώστε από το 2014 να μπορούμε να εκτιμούμε το χρέος συμπεριλαμβάνοντας και το χρέος το οποίο προκαλείται από τα, από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Το ίδιο και για άλλα, εν περιπτώσει, και για άλλους τομείς και για διάφορα άλλα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Θα δείτε ότι στον κατάλογο τον οποίο δημοσιεύσαμε την 23η Απριλίου σας δίνουμε και σε εσά την δυνατότητα όχι μόνο να ε, ελέγξετε τα κριτήρια του Μάστριχτ, έλλειμμα και χρέος, αλλά να πάρετε επίση και συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες θα σας επιτρέψουν να προσαρμόσετε τους υπολογισμούς σας ανάλογα με τις ειδικέ σας ανάγκες, ανάλογα με τα ειδικά σας αιτήματα. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε όλοι πιο φιλόδοξοι, έτσι ώστε να έχουμε και συμπληρωματικές πληροφορίες πέραν των βασικών κριτηρίων του Μάστρικ, που, παραμένουν φυσικά Μίλα με μίλα, τι συγκρίνουμε. Δηλαδή, είναι σαφές ότι στην αγορά εργασίας, δηλαδή στην απασχόληση, αν κοιτάξει κανείς το μητρό των ανέργων με τις στατιστικές για τους ανέργους, καταλήγει σε διαφορετικά στοιχεία, σε διαφορετικούς αριθμούς. Αυτό είναι το κακό. Το καλό βέβαια είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ευρωπαϊκή στατιστική, ε, είναι ο έλεγχος αν θέλετε της, ε, του εργατικού δυναμικού, ο οποίος γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να συγκρίνει τους γερμανικούς κανείς αριθμούς με τους μαλτέζικους, τους κυπριακούς, τους γαλλικούς κτλ για τις εμπορικές συναλλαγές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ενδοκινοτικές. Μέχρι τώρα έχουμε, θα έλεγα, τις λεγόμενες αντικατοπτριζόμενες διαφορές. Πολλές φορές όταν προσθέτει σαν παράδειγμα κανείς τις εξαγωγές από μια χώρα σε μια άλλη, όταν ε, τις ελέγχει σαν εισαγωγές στην άλλη χώρα δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε. Αντιπροσωπεύει το 50% του κόστους γενικά του διοικητικού των στατιστικών ε, δράσεων. Έχουμε προσπαθήσει πολλά να κάνουμε για να μειώσουμε το βάρος αυτό, αλλά μέχρι τώρα δεν το έχουμε πετύχει. Τώρα θα θέλαμε εμείς να ξεκινήσουμε μια νέα ε, πρωτοβουλία η οποία λέγεται SingStat, Single Market Statistics, Θέλουμε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα είδος ε, συμβάσεως Schengen για τα δεδομένα ή ένα cloud Schengen, ένα σύννεφο για τα δεδομένα, όπου οι ρυθμίσεις από τη μία χώρα να μπορούν να εισραίουν χωρίς εμπόδιο στις άλλες χώρες. Και οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνουμε ε, επικεκαλυμμένες μετρήσεις. Εδώ οι χώρες βέβαια θεωρούν ότι απειλούνται ε, ότι θα χάσουν κυριαρχία γιατί πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στους γείτονές τους. Αλλά έτσι μόνο θα μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα το οποίο να μην είναι απλά ε, μία μορφή συντονισμού. Η αλλαγή λοιπόν ε, γίνεται μέσω του ελέγχου, της εποπτείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα υπογεγραμμένα, τις υπογεγραμμένες δηλώσεις ποιότητας, διασφάλισης ποιότητας, Βλέπουμε τι δεν έχει πάει καλά και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες επί παραβάση και αν χρειαστεί να οδηγήσουμε τις χώρες στο δικαστήριο. Αν πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα καταλαβαίνω γιατί προσβλέπετε τόσο πολύ στον τριγωνικό διάλογο για το ΙΣΕ 2010. Ξέρω ότι ο εισηγητής μας δεν είναι ένας εισηγητής ο οποίος ε, είναι άτολμος και συμβαίνει να είμαι εγώ ο εισηγητή. Ο Ούντο είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ και εγώ από τη δική μου πλευρά που ήρθατε ενώπιον μας κύριε Ράντε Μάχερ. Η Επιτροπή μας σας έχει αναφέρει μέσω της Προέδρου μας ότι έχει πάντα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ευρωστάτ, ακόμα και τότε που δεν ήταν στο κέντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολλοί στοιχεία για τους πολιτικούς λήπτες αποφάσεων. Αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι θα αυξηθούν τα καθηγοντά σας, θα αυξηθεί και η πολιτική σημασία της Ευρωστάτ. Και θα ήθελα να συμβάλλω και εγώ στην προβληματική που ξεκινήσατε λέτε ότι εμείς σαν πολιτικοί πρέπει να σας πούμε τι είναι σημαντικό στις στατιστικές. <clears throat> Εγώ νομίζω ότι όταν η Ευρωζώνη ξαναβρει την ισορροπία της, όταν βρούμε μια διέξοδο από την κρίση, θα χρειαστούμε πολύ καλύτερες στατιστικές για τις δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στην Επιτροπή μας που πιστεύουν ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να ονομάσει policy delivery σε καλά ελληνικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταμετρήσουμε καλύτερα. Το IAS 20, 20 είναι ένα συνώνυμο κατά κάποιο τρόπο μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας. Αλλά όταν θέλουμε να έχουμε ένα αγώνα κατά της ε, ανεργίας ή κατά της ένδυας, έχουμε εργαλεία τα οποία θα μας δώσουν μετρήσιμες εικόνες για την κατάσταση που είναι που επικρατεί στα μελη Πόσο αποδίδουν οι διαδικασίες κατάρτισης, πόσο καλή είναι η υγειονομική ε, <clears throat> περίθαλψη, πώς είναι η γενική υγειονομική πολιτική για την πρόληψη της ε, ε, παρουσίας ορισμένων ασθενειών. Τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει και η δυνατότητα να έχουμε αρκετά στοιχεία για να εκτιμούμε αν πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις γιατί λέμε πάρα πολλές φορές ότι θα υπάρξουν ε, αυτόματος κυρώσεις όταν υπάρχουν καθαρά μετρήσιμα σφάλματα. Αλλά είναι έτοιμη η στατιστική, το στατιστικό γραφείο να αναλάβει και τις συνέπειες μιας σκλήρινσης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να δίδει στοιχεία για κυρώσεις ή χρειάζεται μια μεγαλύτερη υποστήριξη από την ευρωπαϊκή πολιτική για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη αξιοπιστία των στοιχείων τους. η απάντησή μου θα ήταν ότι βήμα-βήμα θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα ε, πιστοποιητικών αξιοπιστίας που έχουμε ξεκινήσει για τα δημοσιονομικά στοιχεία. Από το πέσει με σημαντικό στοιχείο τα δημοσιονομικά στοιχεία και είναι αρκετά στεναρό το καθεστώς για την ανάντη πιστοποίηση αξιοπιστίας. Το επόμενο στοιχείο για μας είναι το βαθμολόγιο. Είναι μακροοικονομικό, το μακροοικονομικό βαθμολόγιο. Φυσικά συμπεριλαμβάνει και αυτό ορισμένους δείκτες που θα είναι πιο, δίκτυο, να, πιο δύσκολο να εξασφαλίσουμε την ποιότητά τους. Γιατί η συλλογή των στοιχείων για τα θέματα αυτά δεν περιλαμβάνουν μονάχα το δημόσιο τομέα αλλά και τα νοικοκυριά και γενικά τον ιδιωτικό τομέα. Θα είναι πιο δύσκολο για μας λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δώσουμε μια εξίσου υψηλή πιστοποίηση ποιότητας για αυτά τα θέματα. Ο στόχος μας όμως είναι να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο στίχημα, σύστημα για την ε, πιστοποίηση ποιότητος του βαθμολογίου. Εμείς έχουμε λοιπόν ένα κανονισμό στατιστικού χαρακτήρα και επιπλέον τον κανονισμό 479, ο οποίος καθορίζει τη δομή διακυβέρνησης η οποία εξασφαλίζει την ποιότητα. Το ίδιο θέλουμε να προτείνουμε και για το βαθμολόγιο, τους δείκτες του βαθμολογίου στον επόμενο γύρο. Και μετά όταν έχουμε τους κύριους ενδείκτες για την Ευρώπη 2020, όταν σταθεροποιηθούν αυτοί οι δείκτες, όταν αρχίζουν να χρησιμοποιούνται πλήρως, εγώ είμαι σίγουρος ότι μέσω και της πολιτικής συζήτησης θα μας παροτρύνουν περισσότερο να εξασφαλίσουμε την απόλυτη στεγανότητα και αξιοπιστία αυτών των δικτών. Γιατί ο Τσάρτ Κούτχαρτ είχε πει, έχει είναι ο γνωστό νόμο, ότι από τη στιγμή που χρησιμοποιείται ένα δείκτη για πολιτικού σκοπού, πάβει να είναι καλό δείκτη. <clears throat> Υπάρχει βρόχο ανάδραση. τα στοιχεία για, την, ε, για το δημόσιο έλλειμμα δεν ήταν ενδιαφέροντα παρά μόνο όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται για, την, για τους σκοπούς της του Μάστρικ. Όταν λοιπόν χρησιμοποιήκαν στατιστικές για τη διαδικασία λήψης απόφασης, τότε ο δείκτης αποκτά ενδιαφέρον από πάρα πολλέ πλευρές. Και όλα αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Δεν θέλω να συζητήσω ιδιαίτερα για αυτό το σημείο, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την παρουσία ή την απουσία πόρων. Το θέμα των πόρων δεν είναι θέμα απόλυτης παρουσίας ή απουσίας πόρων, αλλά όλα αυτά με επαναφέρουν στην ευρωπαϊκή λύση αυτή τη στιγμή. Το ευρωπαϊκό σύστημα δουλεύει εν παραλληλία. 27 φορές παράλληλα ε, ξαναεφευρίσκουμε τον τροχό στα κράτη-μέλη και τίθεται πια το ερώτημα κατεπηγόντως για το πώς μπορούμε να έχουμε μια αλλαγή του συστήματος για να απελευθερώσουμε τους απαραίτητους πόρους για τα συστήματα αυτά εξασφάλισης της ποιότητας. Ο Ευχαριστώ κύριε Ραντεμάχερ για την παρουσία σας μεταξύ μας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία από την παρουσίασή σας. Ένα από αυτά που αναφέρατε ήταν το θέμα των ενδεικτών για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δείκτες, το τονίζετε και στην ιστοσελίδα σας και το παρουσιάζετε πλήρως. Επίσης για τους δείκτες του περιβάλλοντος, βλέπω στην ιστοσελίδα σας ότι τελειώνουν τα στοιχεία το 2009. Δεν έχουμε τίποτα για το 2010. Όλες οι άλλες σειρές ενδεκτών προχωρούν λίγο περισσότερο για το περιβάλλον σταματά 2009. Αυτό είναι πολύ δύσκολο εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για χάραξη πολιτικών. Και αν θέλουμε επίσης για τα άλλα στοιχεία να τα χρησιμοποιούμε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ε, εξαμήνου. Πώς μπορείτε λοιπόν να μας βοηθήσετε να έχουμε πιο επικαιροποιημένα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων. Το δεύτερο θέμα αναφερθήκατε στις λεγόμενες contingent liabilities, τις ε, υποχρεώσεις οι οποίες είναι υποεξάρτηση, όπως είναι παραγωγικά τα... οι συντάξεις. Δεν ξέρω λοιπόν πώς, κατά πόσο οι λύσεις που προβλέπονται στο εξάπτυχο, στο six pack, σας δίνουν μια λύση στα θέματα αυτά. Γιατί πολλές φορές υπάρχει το πρόβλημα ότι τα κράτη-μέλη έχουν ορισμένες ε, ε, δαπάνες σε χωριστά λογιστικά βιβλία και τις καλύπτουν με εγγύησεις και μόνο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς θα πώς αντιδράτε στα αυτά τα θέματα. Επίσης στην έκθεσή μας έχει γίνει σαφές ότι εμείς θέλουμε να υπάρξει πιο φιλικός χαρακτήρας προς το χρήστη για τις πληροφορίες αυτές. Να έχουμε παραδείγματος χάρη γραφήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για μια καλύτερη <clears throat> παιδαγωγική διαδικασία και καλύτερη κατάρτιση ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα για το πού βρίσκονται τα πράγματα σε κάθε κράτος μέρος. Ξέρω ότι κάνετε προσπάθειες για τα θέματα αυτά. Εγώ είμαι ενθουσιώδης χρήστης των στοιχείων σας, αλλά θα ήθελα να ξέρω με ποιο τρόπο είσαστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε τις αιτήσει του Κοινοβουλίου για περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ε, διαισθητικό τρόπο αντίληψης αυτών των στοιχείων. η πρώτη ερώτηση για μένα είναι η πιο δύσκολη να βελτιώσει κανείς το επίκαιρο των δεδομένων, ιδιαίτερα των κοινωνικών στοιχείων, που έχουν διαφορετική φύση από ότι οι δείκτες που αφορούν τον οικονομικό αυστηρά κόσμο ή τον χρηματοπιστωτικό. Προφανώς και χρησιμοποιούμε και δείκτες και στα πλαίσια της διαδικασίας πέραν του ΑΕΠ. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο επίκαιροι γίνεται Είμαστε πολύ κοντά και σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί εδώ ίσως δεν είναι μόνο θέμα της Eurostat. Στην πρώτη προσπάθεια που κάνουμε για να γίνουμε πιο επίκαιροι, θα έχουμε ε, στενή συνεργασία με το JRC, σαν παράδειγμα, έτσι ώστε να καλύψουμε το κενό ανάμεσα σε μια στατιστική καταμέτρηση και σε έναν αριθμό πολύ πιο επίκαιρο μέσω ενός μοντέλου το οποίο να συνδέεται ε, με τις στατιστικές μεθόδους. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε ξεκινώντας ένα μοντέλο ε, με ε, λογική πάντα την παρατήρηση, με στατιστικές που να βασίζονται στην παρατήρηση. Πάντως στο παράδειγμα που έχουμε οι στατιστική στις τιμές, ο δείκτης ε, κατανάλωσης σαν παράδειγμα είναι ιδιαίτερα επικαιροποιημένος και έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες να καταστήσουμε ακόμα πιο επικαιροποιημένους και τους α, ε, ε, τρίμηνους λογαριασμούς, τους εθνικούς και προσπαθούμε γενικά να λειτουργήσουμε πολύ καλύτερα και στον τομέα των κοινωνικών στοιχείων. Εδώ εξαιρώ βέβαια το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι αρκετά επικαιροποιημένο, αλλά σε τομείς διανομής δεν είμαστε πάρα πολύ. Κατανομή, συγγνώμη, δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Το EU Silk, σαν παράδειγμα, είναι ε, μια, μια στατιστική προσπάθεια στην οποία δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Στην ενέργεια έχουμε προχωρήσει. Αν δείτε τα δεδομένα για την ενέργεια 2012, δημοσιεύονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Το πρόβλημα είναι ότι με τα απόβλητα σαν παράδειγμα δεν, δεν ακολουθείται η ίδια ταχύτητα. Κατάλαβα αυτό που είπατε, θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε το θέμα αυτό όσο περισσότερο μπορούμε, θα προσπαθήσουμε να φτέσουμε στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και σε συνεργασία με το JRC, με το Κοινό Κέντρο ε, Έρευνας, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά. Σχετικά με το SIXPACK, θα ήθελα εδώ να κάνω μία διάκριση ανάμεσα σε τέσσερα επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία. Καταρχάς, ε, το συνολικό χρέος των δημοσίων επιχειρήσεων. Μετά έχουμε τις υποχρεώσεις στον τομέα της κάλυψης των συντάξεων και έχουμε επίσης και τις έμεσες υποχρεώσεις που είναι καρπός του PPP. Για αυτές τις τέσσερις κατηγορίες στόχος μας Προσπαθούμε γενικά να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο αυτών των στοιχείων έτσι ώστε να έχουμε ένα συνολικότερο πακέτο της δημοσιονομικής κατάστασης στις χώρες μέλη σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε contingent liability. Βέβαια πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας. Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ να δούμε ποιος είναι ο ορισμός ο οποίος δίνεται σε νομικό επίπεδο οι ιδρυτές του ευρώ σαν παράδειγμα όρισαν το βάθος αυτής της ε, διαδικασίας. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε ε, τα χρέη, ουσιαστικά τις υποχρεώσεις καλύτερα και να ελέγξουμε τις υποχρεώσεις και όχι μόνο τα έσοδα. Το θέμα είναι να το κάνουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Είναι δύσκολο να τα ολοκληρώσει αυτά όλα σαν στατιστικά δεδομένα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε σωστά το χρέος γενικά θα πρέπει να ελέγξουμε και τα έσοδα αλλά και τις υποχρεώσεις. Προσπαθούμε λοιπόν όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με καλύτερο τρόπο από ό,τι το κάνουμε τώρα. Αύριο ή μεθαύριο έχουμε μια συνάντηση αν δεν κάνω λάθος. Μας ικανοποιεί το ότι ασχολείστε κι εσείς με τα θέματα αυτά. Είμαστε σε στενή επαφή με πάρα πολλούς χρήστες στα πλαίσια μιας έρευνας ετήσιας σε βάση ετήσια ικανοποίησης. Οι χρήστες είναι αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόσφαση στα δεδομένα, αλλά πράγματι θα μας δώσετε πολύ περισσότερες ιδέες για το τι χρειάζεστε και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για να σας ικανοποιήσουμε. Σοφή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα σύντομο ερώτημα. Στις απαντήσεις σας ήδη, στην παρουσίασή σας, μάλλον ήσασταν πολύ θετικός για όλα όσα έχουν συμφωνηθεί, τους νέους κανόνες και τις νέες δομές, αλλά στις απαντήσεις σας ήσασταν πολύ πιο επιφυλακτικός και σκέφτομαι αυτό που μας είπε ο κύριος Όκρεχον πέρυσι που ήταν μεν ευγενής αλλά πολύ απεσιόδοξος ή και αρνητικός καθαρά ως προς το ρυθμό εφαρμογής όλων των συμπεφωνημένων και της δεοντολογίας. Αφού έχουμε κοινό νόμισμα, πόσο μπορούμε να κατανοήσουμε τις εθνικές ευαισθησίες, παραδόσεις, πρότυπα και αποφάσεις. Καλά είναι και αυτά όσο ο καθένας ασχολείται με τα δικά του, αλλά εδώ έχουμε κοινό νόμισμα. Και άρα ό,τι ανοησία κάνει μια χώρα επηρεάζει και τις άλλες. Πώς συνδυάζονται τα δύο, δηλαδή μερικές χώρες απλώς δεν εφαρμόζουν τα συμπεφωνημένα είτε στη στατιστική είτε, είτε δεν υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία είτε και αναλυθεί και από την άλλη πώς αυτό επηρεάζει τις υπόλοιπες χώρες. Να κοιτάξτε. Κι εγώ ήμουν ευγενή και αισιόδοξο, αυτή είναι η δουλειά μου. Αλλά σας μίλησα και για ορισμένους φραγμούς, εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στην εφαρμογή ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ενωσιακού στατιστικού συστήματος. Ελπίζω η απάντησή μου να ήταν έντιμη. Είπα πού είναι τα μπλοκαρίσματα. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που δεν ισχύει μόνο για τη στατιστική. Πρόκειται για την αλλαγή από ένα συντονισμένο από ένα σύστημα συντονισμού εθνικών συστημάτων σε εθνικό, σε ενωσιακό. Αυτό είναι πόδινο βέβαια και συμφωνώ απόλυτα ότι σε αυτήν τη φάση πρέπει να γίνουν πραγματικές και να εφαρμοστεί επιτέλους το σύστημα που προβλέφθηκε από το 2009 στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, όχι απλό συνδυασμό εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Ανέφερα ήδη τη στατιστική, τα στατιστικά στοιχεία για την ενιαία αγορά. Αν φανταστείτε ότι το ΑΕΠ της Ολλανδίας τώρα υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου, που όμως δεν συμφωνούν με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για καμία άλλη χώρα μέλος καταλαβαίνετε το πρόβλημα γιατί η Ολλανδία θα πει ας πούμε δεν εμπιστευόμαστε τα στοιχεία των άλλων θα τα επεξεργαστούμε μόνοι μας και αυτό συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του στο ΑΕΠ βλέπετε τι γίνεται γίνονται αυτόνομα χωριστά υπολογισμοί του ΑΕΠ χωρίς καμία συνέπεια και συνδυασμό, γιατί χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές ο καθένας. Εμείς θέλουμε να σταματήσει πια αυτό το σύστημα. Δεύτερον, το δημογραφικό. προστιγμήν στιγμήν ανεχόμαστε διαφορετικούς ορισμούς για τον ε, πληθυσμό αλλά οι διαφορές ξεπερνούν και το 10% και αυτό μας ανησυχεί. Τον μόνιμο πληθυσμό μιας χώρας. Έχουμε τους κατοίκους δηλαδή. Έχουμε διατυπώσει προτάσεις και θα σας τις υποβάλουμε για να δηλώσουμε ότι πρέπει ο πληθυσμός να μετριέται με έναν και ενιαίο ορισμό. Θα γίνουν αλλαγές, θα γίνουν. Και τον επόμενο χρόνο θα κάνουμε τη δοκιμή που θα δείξει αν τα κράτη-μέλη δέχονται την αλλαγή προς ευρωπαϊκό ενωσιακό σύστημα. Τα γερμανικά κρατήδια που εκπροσωπούνται στο Bundesrat ήδη αποφάνθηκαν κατά του κανονισμού 223 λέγοντας ότι παραβιάζει την επικουρικότητα και τις δικαιοδοσίες τους. Αυτά αντιμετωπίζουμε δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά Δυστυχώ, για λόγους υγείας δεν ήμουν παρόν στην Επιτροπή μας εδώ και δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις πρόοδου τις οποίες έχετε, έχετε επιτύχει. Έχετε διαβάσει το σημερινό άρθρο του Σπίγκελ όμω για την Ιταλία. Είναι αρκετά λεπτομεριακό και φαίνεται από διάφορες έρευνες Ε, έρευνες που έγιναν από την γερμανική κυβέρνηση πώς έγινε και η διαδικασία ένταξης της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή, στη ζώνη του ευρώ και για τον κάπως άδοξο ρόλο που έπαιξε η Ευρωστάτ στα θέματα αυτά. Βέβαια, αυτό αναφέρεται στο παρελθόν. Θα, παρόλα αυτά θέλω να σας παροτρύνω να το διαβάσετε το άρθρο αυτό. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε από αυτό το άρθρο. Γιατί φαίνεται πως με διάφορα τεχνάσματα δημοσιονομικά η Ιταλία κατάφερε να εκπληρώσει τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Νομισματικής ε, Ένωσης, πούλησε ε, παραδείγματος χάρη ε, αποθέματα και διαθέσιμα της Κεντρικής Τράπεζας για να μειώσει το, το έλλειμμά της χωρίς την έγκριση της ε, Ευρωστάτ αλλά στη συνέχεια παρά το γεγονός ότι δεν πήρε την άδεια της Ευρωστάτ η Ευρωστάτ θεώρησε ότι έχουν πράγματι επιτευχθεί τα κριτήρια της, ε, της δίκης του μάσετ. Βλέπετε λοιπόν ότι εσείς σαν επιστήμονας, σαν ερευνητής, μπορείτε να έχετε μια άποψη, αλλά μετά έρχεται η πολιτική εξουσία και τα τροποποιεί όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ φαίνεται ότι αυτή η συμπεριψη της Ιταλίας στη ζώνη του ευρώ ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνους για τη ζώνη του ευρώ. Τι είναι αυτό το οποίο θα βελτιωθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει περισσότερος εμπεριστατωμένος χαρακτήρας σε εσά, ώστε κάτι σαν γι' αυτό με την ένταξη της Ιταλίας δεν θα μπορέσει να γίνει, να επαναληφθεί στο μέλλον. Και ποιος μας λέει ότι αυτό το οποίο έγινε με την Ιταλία δεν θα είναι αύριο η Πολωνία. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πολλές φορές για πολιτικούς λόγους, για λόγους ευκαιριακού χαρακτήρα γίνονται πράγματα διαφορετικά. Το 1998 παραδείγματος χάρη λάμβανε χώρα η εκλογική αναμέτρηση του Κόλ με τον Σρόντερ και αυτό οδήγησε σε ορισμένες αποφάσεις που ελήφθησαν. Εσείς λοιπόν ως υπεύθυνο της Eurostat τι είδου υποστήριξη χρειάζεται από εμά του πολιτικού ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδου κατά κάποιο τρόπο λαθροχειρίε και παρακάμψει. Θα διαβάσω το άρθρο που μου αναφέρατε στο Spiegel. το κατέβασα ήδη στο iPad μου, αλλά δεν μπόρεσα να το διαβάσω ακόμα. Όλα αυτά αναφέρονται σε μια εποχή στο τέλος της δεκαετίας του 1990 όταν η κατάσταση του Eurostat, η κατάσταση του Eurostat και η πόροι της Eurostat ήταν τελείως διαφορετική. Δεν νομίζω λοιπόν μπορούμε να συγκρίνουμε εκείνη την εποχή με τη σημερινή. Για να σας δώσω ένα δίκτυο για τα θέματα αυτά. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή μάλλον που αναφέρεστε, δεν υπήρχε καν μια μονάδα που ασχολείται με τις οικονομικές στατιστικές. Υπήρχε απλώς ένα τμήμα με δύο ή τρία άτομα που επεξεργαζόταν τέτοιου είδους στατιστικές ε, κρατικών λογαριασμών. Και σας ξαναφέρνω στον, στον νόμο του Goodhart το παράδειγμα αυτό ότι οι δείκτες γίνονται όταν γίνονται ορατοί και περίοπτοι τότε πάβουν να είναι χρήσιμοι. Αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη εφευρετικότητα τότε στα κράτη-μέλη για να δημιουργηθούν ορισμένες κατά κάποιο τρόπο επιρροές στις στατιστικές. Οι δείκτες αυτοί τους επεξεργαζόντουσαν τρία άτομα στη Eurostat Τώρα έχουμε 50 άτομα τα οποία ασχολούνται με τίποτα άλλο εκτός από τις, χρηματο, τις δημοσιονομικές στατιστικές. Έχουμε κάνει πολλές επισκέψεις σε πέντε κράτη-μέλη. Πήγαμε όχι μονάχα στο κεντρικό, στην κεντρική στατιστική υπηρεσία των χωρών αυτών, αλλά πήγαμε και σε περιφερειακά γραφεία, σε δήμους και μέσα σε αυτές τις πέντε χώρες περιλαμβάνεται και η Γερμανία και η Αυστρία. Και νομίζω ότι μετά από όλα αυτά μπορούμε τώρα να δηλώσουμε ότι έχουμε πια ένα κάποιο τρόπο στόκ γνώσεων που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε μια καλύτερη αξιολόγηση των οικονομικών στατιστικών σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάθε φορά που βλέπαμε να παρουσιάζεται ένα σημαντικό κίνδυνο για την ποιότητα των δεδομένων, θα ξεκινήσουμε τη λεγόμενη μεθοδολογική επίσκεψη που είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για μια τέτοια αντιμετώπιση κλιμάκωσης των προβλημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους. Για τα δημοσιονομικά λοιπόν αυτά στοιχεία νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό πλανήτη από αυτά που συνέβαιναν το 1998. Αυτό τώρα το οποίο ελείπει από την πλευρά της Eurostat θα έλεγα και πάλι ότι δεν έχουμε επαρκείς πόρους. πόρους. Και το πρόβλημα είναι η επιρροή και ο ρόλος των συναδέλφων μας στα εθνικά κράτη που θα πρέπει και αυτοί να μπορέσουν να ελέγχουν στο δικό τους περίγυρο αυτά που λαμβάνει εκεί η χώρα. Όλα αυτά όμως είναι τμήμα της πρότασης που έχουμε περιλάβει στην ε, τροποποίηση του κανονισμού για τα στατιστικά στοιχεία. Θα είδατε ότι έχουμε προτείνει να ενισχύσουμε το συντονιστικό ρόλο των Εθνικών Στατιστικών Ινστιτούτων και για μένα αυτό είναι ο ελίπων κρίκος για να μπορέσουν οι συναδελφοί μας σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν ότι οι δικές τους στατιστικές αρχές έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να ελέγχουν τα τεκτενόμενα στη χώρα που βρίσκονται. Ευχαριστώ. Ο Λίαμ. Ευχαριστώ τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, για την Ελλάδα. Το Eurostat γνώριζε τα προβλήματα αξιοπιστίας των αριθμών του ελληνικού χρέους πριν ξεσπάσει η κρίση του χρέους και συγκρίνω με αυτά που είπε ο συνάδελφος για την Ιταλία. Ίσως μου πείτε ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι, αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Δεύτερον, αυτά που είπατε για τους δείκτες που καθοδηγούν την οικονομική πολιτική. Τώρα που συζητούμε τη νέα συνθήκη, το Fiscal Compact, αυτά γίνονται ακόμη και πιο σημαντικά. Πώς υπολογίζεται λοιπόν στο Eurostat τέτοια πράγματα και πώς κρίνεται αυτόν τον δείκτη. Το δομικό χρέος θα εξαρτάται πλέον από το έλλειμμα, το τρέχον έλλειμμα και άρα τότε ό,τι ζητάει η συγκυριακή πολιτική. Τότε τι χρειάζεται ο δείκτης αυτός ως καθοδηγητής οικονομικής πολιτικής εφόσον το δημοσιονομικό εργαλείο έχει εξουδετερωθεί. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τελευταίο ερώτημα που συνεχίζει αυτά που είπαν οι οικολόγοι φίλοι μου εδώ. Στο πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη έχει προταθεί ένας δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, την ποιότητα της ανάπτυξης δηλαδή. Στο Eurostat υπάρχει κάποιος τέτοιος δείκτης. Ξέρω ότι μιλήσατε για περιβαλλοντικούς δείκτες, αλλά υπάρχει ένας δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης ή ανθρώπινος δείκτης ανάπτυξης. Στο... Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη σας ερώτηση, αν ήταν εν γνώση η Eurostat. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στην έκθεση που είχαμε διατυπώσει τον Ιανουάριο του 2010. Εκεί λέγαμε, κοιτάξτε τα τελευταία χρόνια τα ανακοινοθέντα τύπου. Θα δείτε ότι από το 2005 η Eurostat με μία εξαίρεση πάντα εξέφραζε επιφυλάξεις για τα ελληνικά στατιστικά δεδομένα. Πάντα δηλαδή συνοδεύαμε με ένα ερωτηματικό ε, τις ανακοινώσεις ε, για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό επιβεβαιώνει το ότι αμφιβολίες είχαμε. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν προβλήματα. Από την άλλη, ήμασταν λίγο σαν τον εισαγγελέα αν θέλετε, ο οποίος έβλεπε κάποια μηνύματα, κάποιους δείκτες, αλλά δεν ήμασταν ικανοί να αποδείξουμε Είχαμε ζητήσει από τους συναδέλφους μας στην Ελλάδα σε όλες τις ερωτήσεις τις οποίες στέλναμε για τα δεδομένα και εγώ προσωπικά είχα πάει στην Ελλάδα όταν έφτασα στη Eurostat σαν πρώτη αποστολή και τους είπαμε ελέγξατε αυτό, αυτό και αυτό και μας επιβεβαίωσαν γραπτά με υπογραφή του Υπουργού ότι όλα ήταν σε σωστά. Ήταν αντίθετο να αποδείξουμε το αντίθετο. Ήταν αδύνατο να αποδείξουμε το αντίθετο. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε το 2010 μια κάπως ασυνήθιστη διατύπωση. Γιατί είπαμε ότι υπήρξε σκόπιμη παραπληροφόρηση. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε είναι πολύ βαριά έκφραση σε σχέση με αυτά τα οποία συνήθως λέμε. Υπήρξε λοιπόν σκοπιμότητα στην αποστολή λανθασμένων δεδομένων. Σε εκείνη τη φάση, το 2010, δεν είχαμε την δυνατότητα να ανοίξουμε το καπάκι και να δούμε ακριβώς ας πούμε τους συγκεκριμένους ισολογισμούς. Τώρα όμως έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Και ακριβώς από τότε, είδαμε, αφού είδαμε τα λογιστικά βιβλία, μπορούμε ε, να μην έχουμε επιφυλάξεις. Τώρα για τα διαφθορτικά ελλείμματα. Αυτό δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούμε στη στατιστική σαν έννοια. Εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο του ελίματος όπως ακριβώς περιλαμβάνεται στον κανονισμό ΕΖΑ. Για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης σε αιτήσια αλλά και φυσικά τριμηνία βάση. Αυτό σας δείχνει ακριβώς και τι θα έλεγα, τον χαρακτήρα της αλλαγής με ταχύτητα. Τώρα για το HDI, όπως χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο για διάφορους λόγους, κυρίως λόγους κριτικής που έχουν ακουστεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα αξιολόγησης στο HDI, το HDI έτσι και αλλιώ περιλαμβάνει πάρα πολλούς δείκτες οι οποίοι αφορούν τις επίσημες στατιστικές, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Εμείς όμως δεν θεωρούμε ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν 20-25 δείκτες από διαφορετικούς τομείς με ένα πρόγραμμα στάθμισης το οποίο να δίνει ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα σύνθετος δείκτης όπως ονομάζεται και η εσωτερική στάθμιση στο δίκτυο αυτό είναι μια διακανονιστική λειτουργία. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε, και εδώ θα ήθελα να σας συστήσω παρακαλώ να σας παραπέμψω στην ιστοσελίδα μας και να δείτε την έκθεση για την αηφόρο ανάπτυξη της Eurostat και εκεί θα δείτε πραγματικά όλα τα συστατικά της του δίκτυα ανθρώπινης ανάπτυξης τα οποία προσμετρώνται σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους, αναδείκτη κάθε φορά. Και αυτό θα θέλαμε να κάνουμε και για την Ευρώπη 2020, θα θέλαμε να λάβουμε τους δείκτες όπως ακριβώς ορίζονται και θα προσπαθήσουμε να τις βάλουμε στις χρονοσυρές μας και να τις συγκρίνουμε σε σχέση με τις αξίες τις οποίες έχουμε τις στατιστικές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια σύμβολα ας πούμε και για τον καιρό. Λέμε ο ήλιος σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Όταν έχουμε μια στραπή, αυτό σημαίνει ότι ένας δείκτης δεν είναι σωστά ενημερωμένος. Είναι ευανάγνωστη η έκθεση αυτή για την αηφόρο ανάπτυξη και θα καταλάβετε σε ποιους τομείς η Ευρώπη έχει προχωρήσει και σε ποιους τομείς όχι. Τώρα, για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις πολιτικές μας, ήδη από τον επόμενο χρόνο, το 2013, θα βάλουμε και τον δείκτη τον λεγόμενο της προσλαμβανόμενης ευημερίας. Στα πλαίσια της έρευνας EU Silk που αφορά ε, τα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη. Εδώ δεν ζητάμε μόνο συγκεκριμένα δεδομένα, αλλά και κάποια άλλα κριτήρια για την εκπαίδευση, για την υγεία, για την εργασία και θα ρωτάμε από τους πολίτες επίσης τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αξιολογούν την υγεία τους και το περιβάλλον τους κάτω από μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και αυτό θα έλεγα μας οδηγεί σε μια πληρέστερη εικόνα, όχι μόνο επί τη βάση των δεδομένων, αλλά και επί τη βάση των αντιλήψεων και των τρόπων με τον οποίο προσλαμβάνουν οι πολίτες την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας κύριε Ράντερ Μάχερ. Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα. Μία από αυτές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο των στατιστικών στις, στους κανονισμούς μας. Αυτή τη στιγμή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραδείγματο χάρη συζητάτε το θέμα της εξαίρεσης από ορισμένες λογιστικές υποχρέωσεις. Έχετε τη δυνατότητα εσείς ως στατιστική αρχή να αποκτήσετε αυτά τα στατιστικά στοιχεία με άλλους τρόπους. Επίσης, είναι πολλές φορές απαραίτητο να έχουμε σε πραγματικό χρόνο συγκρίσιμες πληροφορίες. Έχουμε για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 μια πρόθεση να συμμετέχουν όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και οι περιφέρειες. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πληροφορίες και για τις περιφέρειες μέσα στην εκπόνηση της, ε, της, ε, των μέτρων για την Ευρώπη 2020. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια διάκριση, αν θέλετε, μεταξύ των δύο ερωτημάτων σας. Καταρχήν για τι περιφέρειε και δεύτερον για τον ε, πολιτικό αντίκτυπο των στατιστικών. Εμείς δεν καταμετράμε ακόμα τον αντίκτυπο των πολιτικών μέτρων. Δεν είναι κάτι το οποίο να είναι τόσο κοντά σε μια έκθεση αντικτύπου. Καμιά φορά ναι. Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται και αυτό σε αυτά που κάνουμε στο φυσιολογικό μας πρόγραμμα. Θα βλέπατε λοιπόν να υπάρχει κάποιος αντίκτυπος σε ορισμένους δείκτες. Δεν υπάρχει όμως μια άμεση σύνδεση που να λέει ορίστε εδώ είναι το άχθος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προέρχεται από την τάδε περιοχή πολιτικής και τώρα αλλάζει η νομοθεσία και βλέπουμε ότι τροποποιεί κάπως αυτό το άχθος. Αυτό θα πρέπει να, να καταμετράτε με ένα μοντέλο πρότυπου κόστους, το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Στην προηγούμενη μου ζωή ως επικεφαλής της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας είχαμε πράγματι μία ε, επεξεργασία αυτού του μοντέλου πρότυπου κόστους και μπορούσα να σας δώσουν τα στοιχεία αυτά στη Γερμανία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στις επίσημες ευρωπαϊκές στατιστικές. Για τις περιφέρειες, βεβαίως, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πάρα πολλούς ε, δείκτες δεν έχει πολύ νόημα να, συγκρίνουμε μια μικρή χώρα, τη Σλοβενία παγωσχάρη, με τη Γαλλία. Ιδίως όταν πρόκειται για κοινωνικές στατιστικές ή στατιστικές αγορά εργασίας. Θα πρέπει να κάνει κανείς μια ε, στατιστική σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό κάνει πιο πολυδάπανη λοιπόν τη στατιστική. Για να έχετε αξιόπιστα στοιχεία για μια περιφέρεια θα πρέπει να έχετε το κατάλληλο δειγματοληπτικό, το κατάλληλο δείγμα, μέγεθος δείγματος στην ίδια την περιφέρεια αυτή. Εμείς κάνουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε τουλάχιστον για τις κοινωνικές στατιστικές και τις στατιστικές περιβάλλοντος θα μπορούμε να κάνουμε μια εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο που θα πλησιάσουν αυτό το οποίο χρειάζεται για να συγκρίνεται παραδείγματο χάρη τη Νότια Ιταλία, το Μεσογειώνο με τη Σλοβενία. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Ράντερ Μάχερ, αγαπητέ Βάλτερ. Ξέρεις φυσικά όπως ε, το είπα και στην αρχή το κοινοβούλιο είναι πάντα στο πλευρό σας. Και όταν εκπροσωπούσατε τη Γερμανία θυμάμαι που κάπου διασταύρωσα το ξύφος με το δικό σας στον τριγωνικό διάλογο. Όλοι μας θέλαμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς καταλήγουμε στα στοιχεία από τις περιφέρειες, όπου είχαμε κάποιες διαφωνίες φυσικά εκείνη την εποχή, αλλά τότε υπήρχε ένα πρόβλημα με τη Γερμανία για να μπορεί κανείς να έχει στοιχεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και φυσικά στο Κοινοβούλιο πάντα συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας για την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους εμείς έχουμε πιέσει το να έχει η Ευρωστάτ περισσότερες εξουσίες. Ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει δυνατό με μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, με διαδικασίες τριλόγου και όχι για να αντιμετωπίσουμε μονάχα κρίσεις όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Συνεχίζουμε λοιπόν να υποστηρίζουμε τη δράση σας, τις ε, στατιστικές σας εκθέσεις και ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο. Δεν θέλω να θέσω κανένα ερώτημα, απλώς να τονίσω ότι σας υποστηρίζουμε απόλυτα για να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία, τα στατιστικά είναι ακριβή και αν τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν την κυριαρχικότητα πάνω στα δεδομένα τους, δεν θα έπρεπε αυτό να σημαίνει ότι μπορούν να έχουν και τη δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια τα κράτη ποια είναι η βαθμολογία που τους δίνουν για τη φερεγγιότητά τους οι αγορές. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε μια, ένα αξιόπιστο πλαίσιο για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συγκρισιμότητα των στοιχείων. Σας ευχαριστούμε, ελπίζουμε ότι θα επανέλθετε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων και έχετε δείξει βέβαια τη σε βάθος γνώση σας όλο το το Τον Ευχαριστώ. Do we Έχουμε άλλα θέματα, όχι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι λοιπόν στις 14 Μαΐου εδώ στις Βρυξέλλες από τις 4 και μισή έως τις 8. Είναι πολύ σημαντική η ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα. Είναι το δίπτυχο για το CRD και επίσης για τις υποθήκες. Όλα αυτά στις 14 Μαΐου από τις 4.30 ως τις 8. Merci.